Liebe Kolleginnen und Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε μόνο μισή ώρα στη διάθεσή μας και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο. Λέγομαι Κωνσταντς Κλέρ, έχω τη μεγάλη τιμή να προεδρεύσω στην αρχή της συνεδρίασης αυτής. Δεν είμαι πιο ηλικιωμένη, αλλά είμαι η πιο παλαιότερη στην υπηρεσία μέλος της Επιτροπής Περιφερειακών Θεμάτων και γι' αυτό είναι μια μεγάλη χαρά και μια μεγάλη τιμή για μένα, τουλάχιστον στην αρχή της νομοθετικής περίοδου, να προεδρεύσω της Επιτροπής μας και να προετοιμάσω το έδαφος για το επόμενο Προεδρείο της Επιτροπής μας. Θα ήθελα τώρα να χρησιμοποιήσω ένα λεπτό για να χαιρετήσω όλους αυτούς που επανήλθαν, που επανεξελέγησαν και που θα εργαστούν και πάλι στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω γνωστά πρόσωπα και πάλι εδώ στην αίθουσα και φυσικά χαίρομαι για όλους αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι είναι ε, νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νέα μέλη της Επιτροπής μας και τα οποία θέλουν να εργαστούν στα θέματα της περιφερειακής πολιτικής μια πολιτική για την οποία μπορεί ο καθένας μπορεί να πει πολλά πράγματα για τη δική μου περιοχή. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι μια μοναδική περιοχή και πιστεύω και εσείς πιστεύετε το ίδιο για τη δική σας περιοχή. Μπορούμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό να προετοιμάσουμε την επόμενη περίοδο 2015-2020 για τη χρηματοδότηση στα περιφερειακά θέματα και να ε, εφαρμόσουμε το πλαίσιο το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Να το εφαρμόσουμε λοιπόν το πλαίσιο αυτό στην πράξη και πιστεύω ότι και μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε αυτό στις ε, συζητήσεις και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας και χαίρομαι θα χαρώ μάλλον πάρα πολύ αν μπορέσουμε να το πράξουμε αυτό με το ίδιο συλλογικό πνεύμα που έχει διαπνεύσει τις εργασίες της Περιφερειακές Επιτροπές στην προηγούμενη θητεία προς όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειών της. Και τώρα θα πρέπει να έρθω στα θέματα της συγκρότησης του Προεδρείου της Επιτροπής μας και κηρύττω την επίσημη έναρξη της συνεδρίασης και θα ήθελα να σας αναφέρω επισήμως ότι ο στόχος αυτής της συνεδρίασης είναι η συγκρότηση σε σώμα του Προεδρείου της Επιτροπής μας με την εκλογή καταρχήν του ή της Προέδρου της Επιτροπής μας και κατά δεύτερο λόγο της εκλογής τεσσάρων αντιπροέδρων βάσει του άρθρου 204 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σειρά είναι των ενεργειών μας. Θα ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο, με την πρόεδρο, μετά τους αντιπρόεδρους κατά σειρά. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω τα άτομα τα οποία δεν είναι τακτικά μέλη ή αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής ε, και εκπροσωπούν κάποιον άλλο να επιβεβαιώσω Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Ρούτικ αντιπροσωπεύει την κυρία Χέιτ, η οποία δεν είναι παρούσα και είναι τακτικό μέλος. Δεν έχω άλλη πληροφορία για αναπλήρωση. Θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν και άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία δεν είναι τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη στην Επιτροπή αυτή αλλά παρόλα αυτά είναι παρόντα σήμερα εδώ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Μπορώ λοιπόν να θεωρήσω ότι μπορούμε με την ε, εξαίρεση ενός μέλους που αναπληρεί κάποιο άλλο να έχουμε την πλήρη σύνθεση της Επιτροπής μας. Ο κ. Σόλμπερ και ο κ. Ζαριλά δεν μπόρεσαν να έλθουν, αλλά και αυτοί εκπροσωπούνται από συναδέλφους. Λοιπόν, να ελέγξουμε κατά πόσο υπάρχει απαρτία, δηλαδή το 1, δέκα, το 1 τέταρτο των μελών της Επιτροπής μας. Ζητώ τη γραμματεία αν αυτό υπάρχει, αν αυτό το ποσοστό υπάρχει. Είναι 11 μέλη το 1 τέταρτο και είναι προφανές ότι είναι 11 μέλη. Είναι διαγυμνού οφθαλμού σαφές ότι είναι παρόντα αυτά τα 11 μέλη τουλάχιστον και γι' αυτό μπορούμε να έρθουμε επιτέλους στην πρώτη εκλογή, την εκλογή του Προέδρου της Προέδρου της Επιτροπής μας και θα ήθελα να ακούσω τις προτάσεις. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω το εξής. Ε, θα ήθελα να σας προτείνω εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων μία υποψηφιότητα για την Προεδρία της Επιτροπής μας και προτείνω συγκεκριμένα την υποψηφιότητα της κυρίας Ίσκρα Μιχαήλωβα εξ ονόματος της Φιλελεύθερης Ομάδος και είμαι σίγουρος ότι είναι μία συνάδελφος η οποία μπορεί να φέρει σε πέρας πλήρως αυτό το έργο διότι έχει μεγάλη πολιτική εμπειρία και η οποία έχει εργαστεί στο Βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε άλλους πολιτικούς και διεθνείς φορείς. Έχει λοιπόν μεγάλη διεθνή εμπειρία και εθνική εμπειρία για τα θέματα αυτά και πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλει τα μάλα στη σωστή λειτουργία της Επιτροπής μας. Γι' αυτό, χωρίς να μακρηγορήσω, <clears throat> νομίζω ότι μπορείτε όλοι να δείτε το βιογραφικό της. Πιστεύω ότι μπορείτε να υποστηρίξετε την κυρία Ισκρα Μιχαήλωβα. Σα ευχαριστώ πολύ, λέγει Προεδρεύουσα. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι. Μπορούμε λοιπόν να ρωτήσουμε την υποψήφια αν είναι έτοιμη να αναλάβει την υποψηφιότητα αυτή, κυρία Μιχαήλοβα. Βεβαίω, λέει η κυρία Μιχαήλοβα. Χαιρόμαστε όλοι πάρα πολύ. Δεν έχω καμία άλλη αίτηση για υποβολή υποψηφιότητα. Κανείς δεν θέλει να ζητήσει την μυστική ψηφοφορία και εφόσον έχουμε μονάχα μία υποψήφια μπορούμε να την εκλέξουμε δια βοής και σας προσκαλώ να το πράξετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Συγχαρώ, την κυρία Μιχαήλοβα για την εκλογή της και φυσικά πρέπει να της δώσω την έδρα της Προέδρου. Σας εύχομαι κάθε δυνατή επιτυχία και καλή συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Συγχρόνως μου αναθέτατε μια μεγάλη ευθύνη. Για μένα αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή που μπορώ να συνεργαστώ μαζί με όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής Περιφερειακής Ανάπτυξης και ναι, βεβαίως και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Να ξέρετε επίσης ότι θα κάνω και ό,τι περνάει από το χέρι μου, ό,τι μπορώ για να ανταποκριθώ στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στη συνέχεια της ημερήσιας διάταξης προκειμένου να εκλέξουμε τα μέλη ε, του Προεδρείου, τους αντιπροέδρους μας δηλαδή. ξέρουμε ποιοι είναι οι αναπληρωματικοί που αντικαθιστούν δηλαδή τα τακτικά μέλη στην ψηφοφορία. Ξέρουμε επίσης ότι έχουμε και απαρτία, σωστά. Το επιβεβαιώνει η γραμματεία. Ζητώ λοιπόν τώρα από τις πολιτικές ομάδες ή από 5% τουλάχιστον των μελών της Επιτροπής αυτής να προτείνουν υποψηφίους, μέλη της Επιτροπής μας δηλαδή, για τις θέσεις των Αντιπρόεδρων. Παρακαλώ. Κυρίε και κύριοι, εξ ονόματος της ΓΚΟΕ NGL για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου ε, προτείνω τον κύριο Γιούνου Σομαρτζή Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για την Επιτροπή μας, γιατί και στην προηγούμενη θητεία ήταν ιδιαίτερα ενεργός σε αυτή την Επιτροπή και εκπροσώπησε την, ε, την γαλλική υπερπόντια περιοχή της Ρεϊνιών και μπορώ και από τη δική μου εμπειρία να πω ότι ήταν πολύ ενεργός και πολύ επιτυχής και είναι μια πολύ καλή επιλογή για μας. Ευχαριστούμε. Αυτή είναι η πρώτη υποψηφιότητα. Για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου της Επιτροπής μας. Συνεχίζουμε με τις υποψηφιότητες ή εκλέγουμε. Α, να ρωτήσω πρώτα. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες παρακαλώ για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου. Όχι. Συνεπώς, εγκρίνεται η υποψηφιότητα αυτή. Διαβοής. Εγκρίνεται ο ορισμός του πρώτου αντιπρόεδρου μας. Παρακαλώ, ελάτε εδώ, στο Προεδρείο. Now I'm asking for the Τώρα περνάμε στις υποψηφιότητες για την θέση του δεύτερου αντιπρόεδρου της Επιτροπής μας. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, επωφελούμε από την ευκαιρία αυτή για να σας συγχαρώ για τα σημαντικά καθήκοντα που αναλαμβάνετε ως ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Νομίζω ότι εδώ εκφράζω και την άποψη ολόκληρης της Επιτροπής αυτής για το γεγονός ότι προσβλέπουμε σε πολύ καλή συνεργασία μαζί σας προκειμένου να προχωρήσουμε στα καθήκοντά μας. Για τη δεύτερη αντιπροεδρία λοιπόν προτείνουμε τον κύριο Στάνισλαφ Πόσακ ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στη Τσεχία και έχει βρεθεί και πολύ κοντά στους πολίτες με τις αρμοδιότητες που είχε εκεί, οπότε τον προτείνουμε για τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου της Επιτροπής μας. Ευχαριστούμε. Υπάρχει καμία άλλη υποψηφιότητα παρακαλώ για τη θέση του Αντιπρόεδρου. Ευχαριστώ. Ναι, θα ήθελα να προτείνω τον Πιλίτεβιτς εκ μέρου της ομάδας του EFDD. Λέει η κυρία Νταμάτο. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να επαναλάβετε το όνομα του υποψηφίου που προτείνετε. Γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για πλήρες μέλος της Επιτροπής μας. Έντεριτς. Köszönöm, elnök asszony, rövid kérdés. Mi alapján fogunk szavazni? Főleg... Θέλω να υποβάλω μια ερώτηση παρακαλώ. Πώς θα ψηφίσουμε Έχουμε κάποιο βιογραφικό. Πού θα βασιστούμε. Θα ακούσουμε απλώ ένα όνομα και μετά θα ψηφίσουμε για ένα όνομα απλώ. Ή θα ξέρουμε κάτι παραπάνω. Στο όνομα της δημοκρατίας λοιπόν ρωτάω βάσει τίνος πράγματος ψηφίζουμε. Κανείς δεν μας συστήθηκε και εμείς είμαστε καινούργιες στην Επιτροπή αυτή και στο Κοινοβούλιο οι περισσότεροι, οπότε δεν ξέρω σε τι βάση, που θα βασιστούμε για να ψηφίσουμε για τις θέσεις αυτές της Αντιπροεδρίας. Πρόεδρος, κάθε μέλος της Επιτροπής αυτής μπορεί να προτείνει Αντιπρόεδρο για την Επιτροπή μας, εφόσον τον ε, στηρίζουν κάποιες πολιτικές ομάδες, μια πολιτική ομάδα τουλάχιστον. Ο αντιπρόεδρος έχει δικαίωμα, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος, να παρουσιαστεί. Τώρα γνωρίζουμε τα ονόματα των δύο υποψηφιότητων που έχουμε. Η πρώτη παρουσιάστηκε, η υποψηφιότητα, και η δεύτερη παρουσιάστηκε απλώς με όνομα. Μόνο το όνομα προτάθηκε. Ίσως ε, μπορείτε εσείς να μας πείτε περισσότερα πράγματα για την υποψηφιότητα αυτή και μετά θα σας εξηγήσω βάσει ποιας τεχνολογίας θα ψηφίσουμε για τις δύο αυτές υποψηφιότητες. Παρακαλώ, κύριε Μάτο. Πέραν του ότι θεωρώ ότι δεν γνωρίζουν όλοι τα βιογραφικά όλων των υποψηφίων, θεωρώ ότι η αιτιολόγηση της υποψηφιότητας ε, του ε, υποψηφίου ε, οφείλεται στην αρχή της δημοκρατίας, να τηρούμε λοιπόν τους, την δημοκρατικό χαρακτήρα του να μπορούν να είναι παρόντες σε, όλες τα, όλα τα προεδρία, άρα να υπάρχει η παρουσία και του FDP. Thank Ευχαριστούμε. Αυτή λοιπόν ήταν η παρουσίαση της νέας υποψηφιότητας. Έχουμε λοιπόν δύο υποψηφιότητες. για την δεύτερη θέση προεδρία. Πρέπει εδώ να σας πω επίσης ότι σε αυτή την περίπτωση η ψηφοφορία θα γίνει μυστικά, δεδομένου ότι υπάρχουν δύο υποψήφοι. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα σε μία ψήφο. 13 ψήφους έχει το ΕΛΚ, 12 οι σοσιαλιστές, το ECR έχει 3 ψήφους, η ΑΛΔΕ 4 ψήφους, η ΓΚΟΕ 3, η Πράσινη 2, το EFDD 3 ψήφους και η μη γεγραμμένη 3. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στον πρώτο γύρο κερδίζει ο υποψήφιος ο οποίος έχει μπορέσει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ε, ψήφων. Στις ψήφους συμπεριλαμβάνονται οι ψήφοι υπέρ του υποψηφίου, του ενός ή του άλλου. Εντάξει, θέλω επίσης να σας ενημερώσω για το ότι θα ψηφίσουμε με μυστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Συνεπώς, πρέπει να ξέρουμε, έχετε όλοι τις κάρτες σας για να ψηφίσετε. Έχετε τις κάρτες σας. Ευχαριστώ. Ενθαρρυντικό. Μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε. Έχουμε λοιπόν δύο ονόματα. Έτεριτς, είναι ο κύριος Έτεριτς, ένας υποψήφιος. Και ο κύριος Πόλτσακ είναι ο δεύτερος υποψήφιος. Α, όχι, ο πρώτος είναι ο κύριος Πόλτσακ. Ναι, γιατί ήταν ο πρώτος που προτάθηκε. Σας ευχαριστώ για τη διόρθωση αυτή. Σας ευχαριστώ. Um, so we Έχουμε λοιπόν τα ονόματα. Η σειρά τώρα των υποψηφίων θα είναι αλφαβητική. Γι' αυτό και πατώντας το πράσινο κουμπί ψηφίζουμε για τον κύριο Έτεριτς και με το κόκκινο κουμπί ψηφίζουμε για τον κύριο Πόντζακ. Το άσπρο κουμπί σημαίνει αποχή. Αν κάνετε λάθος κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί που επιθυμείτε κατά τη διάρκεια που ισχύει ακόμα η ψηφοφορία που δεν έχει κλείσει ακόμα δηλαδή, και τότε αλλάζετε την επιλογή σας. Έτσι, τι ρωτάτε για το λάθος, αν κάνω λάθος. Επαναλαμβάνω, πράσινο κουμπί για τον κύριο Έτεριτς και κόκκινο κουμπί για τον κύριο Πόλτσακ. Είμαστε έτοιμοι. εκτός μικροφώνου παρεμβάσεις για το πόσο δουλεύουν τα μηχανήματα ή όχι. Πρόεδρος, δεν ξέρω πώς να το ελέγξω. Δεν έχουμε εδώ στην αίθουσα κατάλογο με τους ε, τραγουδιστές της όπερας όπως είχαμε στην Ολομέλεια για να κάνουμε τη δοκιμαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίστε παρακαλώ. Uh, are you ready? Okay. I close the Πέρας της ψηφοφορίας, εφόσον έχετε ψηφίσει όλοι. Αποτελέσματα. 39 ψήφισαν, λέει η πρόεδρος. 3 πάτησαν το πράσινο κουμπί. 30 πάτησαν το κόκκινο κουμπί. Και 3 ψήφισαν αποχή. 36 είναι οι καταγεγραμμένες ψήφοι που είχαμε. Ο κύριος Πόλτσεκ λοιπόν εκλέγεται στη θέση του δεύτερου αντιπρόεδρου. Έλατε να καθίσετε εδώ δίπλα μας παρακαλώ. Η γραμματεία με ενημέρωσε πως ε, έκανα ένα σφάλμα όταν είπα ότι θα πρέπει να ελέγξουμε το σύστημα. Και ίσως ε, ορισμένοι εξημών μπορεί αμφισβητήσετε το αποτέλεσμα των, της εκλογής. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ να επαναλάβουμε. Δεν πρόκειται για δοκιμή, για τεστ, πρόκειται για πραγματική εκλογή του δεύτερου αντιπροέδρου. Ευχαριστώ λοιπόν για τις παρατηρήσεις σας, για να είμαστε σίγουροι ότι η εκλογή πήγε καλά, θα πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. την ψηφοφορία για τον δεύτερο αντιπρόεδρο με πράσινο ή με κόκκινο κουμπάκι. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Και επαναλαμβάνω αυτά που μόλις μου είπαν. Ο κύριος Πότζακ είναι το πράσινο κουμπί και ο κύριος Κέροτζ με το, σύγουρο, με το πράσινο ο κύριος και ο κύριος Πότζακ με το κόκκινο. No, you can, you can no, you should not. Okay, everybody, everybody voted. So, thank you. Ψήφισαν άπαντες. Ωραία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. 38 εψήφισαν. 2 ψήφισαν αποχή. Έχουμε λοιπόν 38 ψήφους. 4 πήραν το πράσινο και 30 με το πήραν κόκκινο. Επιβεβαιώνεται πάλι το αποτέλεσμα και βρίσκεστε στην σωστή θέση. Συγχαρητήρια. I hope the Ελπίζω πως, με την... πως την τρίτη φορά θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να ακούσουμε ψηφιότητες και να αποφασίσουμε. Παρακαλώ το όνομα του τρίτου αντιπροέδρου από, πρόκειται από το ΕΛΚΟ Γιώργιν Τζέλερ, ένας από τους συγητές μας στην προηγούμενη θητεία και είναι πρόσωπο με ιδιαίτερη ε, πείρα πάνω στο θέμα. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Okay. Are there other Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητε. Παρακαλώ. Ομάδα EFDD, Ρόζα Ντεμάτο. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή της ομάδας μου και ευχαρίστως ε, να σας ε, βοηθήσουμε όπου θελήσετε κάποια βοήθεια για την διεξαγωγή ψηφοφοριών. Ευχαριστώ. Thank you very much for this declaration. It means that you... Ευχαριστώ. Άρα δεν έχετε κάποιον υποψήφιο. Έχετε. Ρόζα Ντεμάτο. So, other nominations? Άλλες υποψηφιότητες. Λοιπόν, Έχουμε δύο υποψηφίους. Θα επαναλάβουμε την άσκηση που κάναμε προηγουμένως με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για να κατανείμουμε τα χρώματα. Η κυρία Νταμάτο είναι πράσινη. κύριος Τσέλερ θα είναι κόκκινος. Είναι σαφές σε όλους. Πάμε, ψηφίζουμε. Now I close ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα θα ανακοινώσω τώρα. 39 ψήφισαν. Δύο αποχές. Τρεις ψήφους για την κυρία Νταμάτο και 34 ψήφους για τον κύριο Τσέλερ. Προσκαλώ, λοιπόν, τον κύριο Τσέλερ να έλθει στο Πρόεδριο εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν για τη θέση του τέταρτου αντιπρόεδρου. Ναι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω από την πλευρά της Σοσιαλιστικής Ομάδος να προτείνω τον Ιταλό συνάδελφό μας Ανδρέα Κοσολίνο, ο οποίος ήδη ήταν παρόν στην προηγούμενη θητεία στην Επιτροπή μας, ιδιαίτερα επιτυχώς, και ελπίζω ότι θα μπορέσει να αποβεί ένας πολύ καλός αντιπρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Σας ευχαριστώ. Άλλες προτάσεις. Παρακαλώ. Για τον ίδιο λόγο προτείνω τον Bill από την FDP. Ευχαριστώ. Σε Εάν το επιτρέπει ο κανονισμό, τότε το ζητώ. Από ό,τι γνωρίζω, επιτρέπεται. Έχουμε δύο λοιπόν υποψηφιότητε για την τέταρτη θέση αντιπροέδρου. κύριος Γκοζολίνο, είναι η πρώτη πρόταση. Και η δεύτερη για τον κύριο Έτεριτς. Παρακαλώ. Κύριος Μποστινάρου. Από ό,τι ξέρω κυρία Πρόεδρε, το όνομα το οποίο γνωρίζω είχε τεθεί σε υποψηφιότητα και καταψηφίστηκε. Γιατί να συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε αυτή την ενέργεια όταν ένας υποψήφιος έχει απορριφθεί από μεγάλη πλειοψηφία της Επιτροπής μας. Ποια είναι η λογική. Μας επιτρέπουν οι κανονισμοί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Γιατί το ίδιο όνομα ήταν υποψήφια στο παρελθόν και καταψηφίστηκε. Θέλετε να το κάνουμε στο δίνεκες. Κατανοώ αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς οι κανονισμοί από ό,τι γνωρίζω δεν λένε τίποτα σε σχέση με την επανάληψη της πρότασης υποψηφιότητας. Έχουμε διαφορετικές θέσεις και έχουμε διαφορετικές υποψηφιότητες. Οι συνάδελφοι έχουν θέση ως υποψήφιο το ίδιο άτομο, έχει κάθε δικαίωμα να είναι υποψήφιος. Σας προσκαλώ λοιπόν να ψηφίσετε για την τέταρτη θέση αντιπροέδρου. Πράσινο σε αυτήν την περίπτωση για τον κύριο Κοτσολίνο. Κοτσολίνο. Κοτσολίνο. Και το κόκκινο για την κυρία, για τον κύριο Έτεριτς. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Are ready? Είμαστε έτοιμοι. Πέρας στις ψηφοφορίες Να δούμε τα αποτελέσματα. Mm-hmm. We have 37 votes. 37 εψήφισαν. Μία αποχής. 32 υπέρ του κυρίου Κοτσολίνου και 4 υπέρ του κυρίου Έθεριξου. Κύριε Κοτσολίνο, σας προσκαλώ να έρθετε στο Προεδρείο. Um, with this final step... Και τώρα έχουμε περατώσει τη διαδικασία συγκρότησης του Προεδρείου της Επιτροπής μας και η τελευταία μου πληροφόρηση προς ε, εμάς είναι ότι θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η πρώτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής μας Περιφερειακών Θεμάτων θα λάβει χώρα στις 23 Ιουλίου από τις 3 έως τις 6.30 το απόγευμα επίσης στις 24 του μηνός από τις 9 έως τις 12.30 το πρωί στις Βρυξέλλες. Θα σας δώσουμε στοιχεία για την, ομα... για την αίθουσα το ταχύτερο δυνατό. Σας ευχαριστώ και γεια σας.